Welcome Καλώς ορίστε. Παρακαλώ θα απαιτηθεί πολύς χρόνος. Γι' αυτό ξεκινάμε. Um, uh, uh, λοιπόν, μπορούμε παρακαλώ να αποδεχθούμε την ημερήσια διάταξη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σημείο 2. Ε, όλες οι γλώσσες είναι διαθέσιμες εκτός από τα μαλτέζικα, κροατικά και γοηδελικά. Να πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα υποδεχθούμε και τους υπεύθυνους από μια περιοχή της Γαλλίας που ασχολούνται με θέματα απασχόλησης των νέων. Τους έχει προσκαλέσει ο κύριος Λοϊαρίκα. Ίσως έρθουν αργότερα και δεν θα είναι εδώ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Κάτι καλό και για αυτούς και για μας. Λοιπόν, εγκρίνουμε και τα πρακτικά του μηνός Μαΐου και θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. και αν είναι απαραίτητο θα κάνουμε και κάποιο διάλειμμα, αλλά ξεκινήσουμε να δούμε πού θα φτάσουμε. Ξεκινάμε με την γνωμοδότηση για τη εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας για την εσωτερική αγορά με την Ελβετία. Συμβιβαστική α, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική B. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική C. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική D. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική E. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θα ψηφίσουμε τώρα για το σύνολο όπως τροπολογήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ. Okay, Θα ψηφίσουμε τώρα για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 163. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία, ή μάλλον συμβιβαστική AP υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική L. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 179. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική M. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 185 υπέρ κατά αποχές δεκτή 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την 195 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή ε, Next one. That was amendment 196. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική O υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέτζι 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέτζι 26 κατά διέρεση ψήφος πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική πι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική PB υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική AI υπέρ κατά αποχές δεκτή 223. ή Α, για μια στιγμή. 223 και 224 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθησαν. Συμβιβαστική PA υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 232 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για τη 232. Ψηφίζουμε. Πέρασε οι ψηφοφορίες. Απερίφθη. Με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 233. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική QA υπέρ κατά αποχές δεκτή. 238 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 237 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 239 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 240 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.46 με προφορική τροπολογία από τον Σον Σάιμον μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ρέτζι 31 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την Ρέτζι 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη. 247 τώρα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 248 με προφορική. Αντικαθιστούμε το avoid από το overcome υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Και μετά έχουμε την τροπολογία 6. Έχει αποσυρθεί η 6. Η 6 έχει αποσυρθεί και αντικαθίσταται από μια προφορική του κυρίου Μπέκερ. Διαβάζω την προφορική. Στο 12α. Η πολιτική της αγοράς εργασίας είναι εθνική αρμοδιότητα που συντονίζεται και υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το τι με τη συνθήκη και τα μέτρα στήριξης της κινητικότητας θα πρέπει να είναι συμβατά με τις βασικές αρχές της συνθήκης, ιδιαίτερα την ισότιμη αντιμετώπιση και τις ε, ε, αντίστοιχες δίκαιες αμοιβέ. Εντάξει κύριε Μπέκερ αυτό ήταν. Το διαβάσατε πάρα πολύ ωραία λέει ο κύριος Μπέκερ. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία Μπέκερ. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Ρέγγι 32 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2.52. Ποιοι είναι υπέρ, Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.54. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Τρεις ψήφοι διαφορά. Υπέρ έγινε δεκτή. 2.55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. 31 υπέρ 22 κατά. Λοιπόν, 2.56 υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.57 υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική QB υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. 260 υπέρ κατά. Αποχές. Απερίφθη. 261 υπέρ κατά αποχές δεκτή 262 υπέρ κατά αποχές δεκτή 263 υπέρ κατά αποχές δεκτή 264 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ρέτζι 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 265 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 266 υπέρ κατά αποχές δεκτή 268 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 268. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη. Λοιπόν, Ρέτζι 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.73 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 2.75 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Έλεγχος για την 2.75 ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 41 ψήφοι υπέρ. Συμβιβαστική τι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 288. Τέλος. Δεκτή. 289. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 290. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 291 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 292 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική U υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πάμε στη σελίδα 15 τώρα. 329. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέτζι 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική VA υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική Y υπέρ. Στη σελίδα 17 λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, συμβιβαστική Y υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική WA υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη σελίδα 19, συμβιβαστική 370 ή μάλλον τροπολογία 370 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική X υπέρ κατά αποχές δεκτή. την 20 τώρα. 380 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 382 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 384, 385, 386, 387 388 και 389 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 390 και 392 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απερίθησαν. 393 υπέρ, κατά, αποχές, απερίθη. 394 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Περνάμε μετά στην 395 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 398 μαζί με τη συμβιβαστική Z 398 με Z υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 22 συμβιβαστική AA. Ποιοι είναι υπέρ της AA κατά αποχές δεκτή. Έχω μετά την προφορική τροπολογία στο 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 4-15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4-15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες δεκτή. 25 υπέρ 22 κατά. Λοιπόν, 20, 17, 4, 18 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. Θέλετε να υπάρξει έλεγχος λοιπόν για την 20 και τα λοιπά. γίνεται δεκτή. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τέσσερα εικοσιτρία υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 424 εικοσιτέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4.25 ή μάλλον 21. Ποιοι είναι υπέρ της 21. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 427 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 426 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 429 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 και 430 μαζί υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 22 και 430 από κοινού άρχεται η ψηφοφορία Πέρα της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Τέσσερα 4-31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 23 και 4.32 μαζί. Και 4.33 υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 433, 432 και 23 από κοινού. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική AB. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 442 υπέρ. Κατά αποχές, Απερίφη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 442. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 443 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ρέτζι 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 447 υπέρ κατά αποχές απερίφη συμβιβαστική AC υπέρ κατά αποχές δεκτή 451 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απερίφη Συμβιβαστική AD υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην 26 και στην 460 και είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 461 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική AE υπέρ ΑΕ, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 27 τώρα. 479, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, για την 479 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της οφορία εγκρίθηκε. Με δύο ψήφους διαφορά. 480 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 480. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίθηκε. 13 ψήφοι διαφορά. AF συμβιβαστική τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 485 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 485 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Ρέγγι 58. Στη σελίδα 28. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 487. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπάρχει τώρα μία προφορική τροπολογία στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του εισηγητή. Τα μέλη γιούρες και γιούρες εταίροι Μπορούν επίση, ε, μάλλον εφαρμόζεται και σε αυτού, οι αρχέ κτλ. Υπέρ παρακαλώ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 490. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 492. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Ρέγγι 59. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AG. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 497. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική AQ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 30 τώρα. Συμβαστική AH υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5.19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 520 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 522 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 523 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 525 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 525. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της οφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 527 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 528 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 529. 530, 531, 532 και 533 είναι ταυτόσιμες Τις ψηφίζουμε μαζί λοιπόν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 536. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 538. 538. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 500. 539 και 540 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 542 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 544 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 544. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 545. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 547. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 548. Όχι, καταπίπτει. Τροπολογία 549. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 550 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 551 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 30 και ρέγγι 62. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 557 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AJ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. Τροπολογία 33. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 562, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 563, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 564, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για την 564. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της οφορίας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Τροπολογία 565 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε και για την 565. Ηλεκτρονικά μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Συμβιβαστική ΑΚ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 567. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 568 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 568. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες, Απορρίφθηκε. Τροπολογία 569 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 573. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 574. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 574 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της φοφορίας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 575 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 576 υπέρ, κατά, αποχές, 575 λέει πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 576 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 577 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 578 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 579 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 580 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 581 υπέρ κατά Εδώ έπρεπε να έχει συν στο κατάλογο ψηφοφορίας και όχι... Λοιπόν, ξανά. τροπολογία 581. Ψηφίζουμε και πάλι. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική AL. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 586. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 587. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 588. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AR υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα, στη σελίδα 36, συμβαστική AM υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39. με την 618, 619, 620, 621, 622 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 625. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 626. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 627 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 628 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 629 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 630 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 631 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καλά. Θα ελέγξουμε την 631 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη Εγκρίθηκε. Ρέγγι 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 632. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 634. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε. 634. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις 634. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 635. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 636. Α, να ελέγξουμε για την 635. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε. Μπορείτε να ψηφίσετε ακόμα. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 636. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 636. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 637. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. 637. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 638 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 640. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 640 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα τη σοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 641. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική AN. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 648 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 648. Πέρας της βοβορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 649 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 650 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 650. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας τις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 651 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Απορρίπτεται θέλω να πω. Απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 653 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 654 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 655 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 656 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 656. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 657. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 72. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 658. Υπέρ, όχι, καταπίπτει αυτή, δεν την ψηφίζουμε. Και πάμε στην τροπολογία 659 και 660 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 661. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγξουμε. 661. Ψηφίστε. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 662. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 663. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 664. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 665. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 666 προφορική τροπολογία του εισηγητή για τα μέλη και τους εταίρους γιούρες. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 667. Προφορική τροπολογία του εισηγητή για κάθε Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού που πρέπει να καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών λαμβάνοντας υπόψη Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Όχι. Όχι. Ρέγγι 75 πάμε τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 673 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 675. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 676. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 677 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 670... Α, να ελέγξουμε. 677. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 678. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 678. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της φοφορίας, εγκρίθηκε. Με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 680 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 681 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 682 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 683 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 684 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 689, 690 και 690 διακόπτη πρόεδρος. Α, κύριε Λένερς, συγγνώμη, αλλά η πρότασή μου για διαγραφή αφορά τις κατεξουσδότηση πράξεις, αλλά Καλύτερα λοιπόν θα ήταν να αποσυρθεί η τροπολογία μου αυτή. Καλώς κύριε Λένες. 689 και 691 τα ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 692. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 693 καταπίπτει. Πάμε στην 699 κατευθείαν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική A, α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία στην επόμενη σελίδα, 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική B, β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική σί. γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία. Θέλει κάποιος να ελέγξουμε την 68. Ναι, ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε 68. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρίτζι 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε ή στη σελίδα 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 82 και 83 και 84 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική FA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 100. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της Απορίθηκε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Όχι, 106. 106. Κατά τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 106 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Α, Δεύτερο τμήμα τώρα της 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. 109. Μπορείτε να ψηφίσετε. Απορρίφθηκε. 110. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 112. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 113. Υπέρ, κατά, αποχές Απορρίφθηκε. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 124 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 14 υπέρ, α όχι, καταπίπτει αυτή. Οπότε πηγαίνουμε στη συμβαστική H, ήτα, H, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 49, τροπολογία 134, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 135. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 και 138 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α, Ιώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, Ιώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 153, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 17, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 156 με την 158 μαζί υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 161 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη έκθεση γνωμοδότηση μάλλον. Στην τροποποιημένη γνωμοδότηση λοιπόν, ηλεκτρονικά, πέρα στις ψηφοφορίες, 44 ψήφοι υπέρ και 5 κατά. Ευχαριστούμε κύριε Μπέκερ. Αλλά δεν τελειώσαμε μια στιγμή πρέπει να ψηφίσουμε και το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου, το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου, ονομαστική ψηφοφορία, όπως πάντα. Συνεπώς, ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 44 ψήφοι υπέρ και 5 κατά. Ε, το αποτέλεσμα λοιπόν θα ψηφιστεί και θα συμμεριληφθεί στην τελική έκθεση. Αν το ζητήσουν, το 1 τρίτο των βουλευτών που παρίστανται. Ως εκ λοιπόν σας ε, ζητώ να μου πείτε αν θέλετε να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα της συμφορίας στην έκθεση, όχι μόνο στα πρακτικά δηλαδή, αλλά και στην έκθεση. Ναι, μάλιστα, ωραία λοιπόν. Η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε και τον κύριο Μπέκερ. Και έχουμε και άλλες συμφορίες. Ναι, ναι. Κύριος Μπέκερ, να μας πει αν ε, έχει κάποιο σχόλιο για την ε, έκθεση αυτή. Σχετικά με την εντολή του για την ε, έκθεση αυτή. Να ψηφίσουμε λοιπόν και το θέμα αυτό. Για το κατά πόσον θέλουμε να δώσουμε την εντολή αυτή στον εισηγητή. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Όλοι ψηφίσατε σε σχέση με την εντολή. Προς τον κύριο Μπέκερ. 28 ψήφοι χρειάζονται, έχουν ψηφίσει όλοι. Μάλιστα, όλα ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία. 42 λάβατε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο. we go to uh, the vote. Μάλιστα, τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεση για την δημιουργία μια ανταγωνιστική αγορά εργασία για τον 21ο αιώνα, αντιστοίχηση δεξιοτήτων και προσόντων, με τη ζήτηση και τι ευκαιρίε απασχόληση ω τρόπο ανάκαμψη από την κρίση. Έτοιμοι για τη νέα ψηφοφορία. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 έχει καταπέσει ή όχι. Θα την ψηφίσουμε την 33 ως προσθήκη στη συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. να κάνουμε έλεγχο της ψηφοφορίας αυτής, έναρξη ψηφοφορίας. Δεν έχει κλείσει ακόμη ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. τώρα να ψηφίσουμε 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 35. Δεν έχει κλείσει ακόμα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 37 αποτελεί προσθέκη στην συμβαστική Β, το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική C, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Για τη συμβιβαστική C. Ενάξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Στη σελίδα 5, η 52, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 54 μαζί με την 55, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 69, να ελέγξουμε παρακαλώ, η ηλεκτρονικά στην 69. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 71. Πέρα ψηφορίας. Εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ. Να συμμετάχετε όλοι στη ψηφοφορία. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η E. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 66. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχος για την 66. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε και μία προσθήκη στη συμβιβαστική F στο δεύτερο τμήμα. καλή τα κράτη-μέλη with care responsibilities. Με ευθύνε λέξεις. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Ας το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. Και είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία, δεν έχει ολοκληρωθεί. 28. Uh, then we it's closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική δί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογία ή 90. 91, 92, 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Η 95. Καταπίπτει. Η 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 98 με μια προφορική τροπολογία της ε, Άλντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφεται. Η 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Επιτροπής υπο, προ, 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 101 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 102 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Σελβαστική Ι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AIDS. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζητείτε έλεγχος για την 111. Έναρξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 ψήφοι υπέρ. Και 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 113. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, Επιτροπής Πολιτισμού 5 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 6 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συνδαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 110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 κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική μη. Μ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Επιτροπής Πολιτισμού 8. Στη σελίδα 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Επιτροπής Πολιτισμού 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική εν, νη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 164, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται πολιτισμού 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173. Υπέρ. Πρώτο τμήμα μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183. Ναι, and what? Yeah, we Yes, we'll vote on Amendment 183. Την 153 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 181, συγγνώμη. Πέρα της Φορειάς, Εγκρίνεται. 192. Σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται συγγνώμη, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 192. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο, τρίτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193. Υπέρ. Καταπίπτει, καταπίπτει 193. Πολιτισμό 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 194. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 195. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται του πολιτισμού 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 9 του πολιτισμού, του υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 204. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ταφ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206, υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η Επιτροπή Προπολογισμού. Καταπίπτει. Η Επιτροπή Προπολογισμού 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τη Επιτροπή Προπολογισμού η τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R. Υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Επιτροπή Προπολογισμού 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Επιτροπή Προπολογισμού. Πολιτισμού. Με προφορική τροπολογία της Άλντε. Για να αλλάξει η λέξη revision σε review. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 16 τη Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή. Α, συμβαστική W. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 228. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 228 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Η 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε και την 229. Πέρας ψηφοφορίας. Η 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 235 υπέρ Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η 236 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 237. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική χ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 243 προσθήκη Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. 246. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 247. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Υψηλόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 249 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 252. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβιβαστική ζήτα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Πολιτισμού 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Πολιτισμού 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Πολιτισμού 30. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 258 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 259 και η 260 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε παρακαλώ την 259 και 260. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Η αλφα-αλφα. συμβαστική Υπέρ. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Όχι. να το ελέγξουμε παρακαλώ, γιατί δεν ήταν σαφές. Πέρασε. Να ψηφίσουμε κάθε μία λοιπόν ξεχωριστά. Αφού έχουμε ισοψηφία. Δύο εξένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος, βέβαια. Ψηφίζουμε ακόμα ηλεκτρονικά την 261. Εγκρίνεται. 262, 263, 264 καταπίπτουν. Α, τη 264 δεν ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 265. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266. Υπέρ. Καταπίπτει και 267. Πολύ ωραία. Η 267. Ψηφίζουμε την 267 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αλφαβήτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 270. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιτροπής Πολιτισμού η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την συμβαστική AC έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Ισοψηφία. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν όλες τις τροπολογίες. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 273 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 273. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 273. Για την 273. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 274 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει, καταπίπτει 276, συγγνώμη λέει πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 277. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 278. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 279. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 327. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ψηφίζουμε τώρα την 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική AD. Υπέρ. Κα, υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβαστική αλφα αλφα ε, μάλλον. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 297 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η Επιτροπή Πολιτισμού 20, όχι. 298 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται ή 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Η 303 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Η 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Επιτροπής Πολιτισμού 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επιτροπής Πολιτισμού 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική AF Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 307. Πέρα στις ψηφοφορίες δεκτή. Συμβιβαστική AF, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. AH, συμβιβαστική ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την AH. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες δεκτή. Φτάσαμε στην 317. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.18 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. AI ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. AP Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 329. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AJ Προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην 339 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 340 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 341 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 342 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AK υπέρ. Κατά. Δεκτή. 347 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 348 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AL υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AM υπέρ κατά αποχές δεκτή. 358 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική AN υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική AO υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή Δέκα υπέρ κατά αποχές απερίφθη Έντεκα υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές δεκτή Δεκατρία υπέρ κατά αποχές, απερίφθη. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 16 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 16. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη. 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές ε, α, συγγνώμη, έχει καταπέσει 19. Περνάμε τώρα στην 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές απερίφη 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τελική ψήφος τώρα, όπως τροπολογήθηκε. Πέρας της ψηφοφορίας 27 υπέρ 13 κατά. Το αποτέλεσμα της ονομαστικής συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον ζητηθεί από το 1 τρίτο των βουλευτών. Όσοι ψηφίσατε λοιπόν θέλετε να συμπεριληφθεί. Υπάρχει το 1 τρίτο με το χέρι σας διανατάσεως χειρός. Πράγματι το 1 τρίτο το επιθυμεί. Θέλετε κάποιο διάλειμμα. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Yes. <clears throat> Okay, friends, we'll try to finish. Ah. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε. Θα μας χρειαστεί ίσω λίγο παραπάνω χρόνος. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κύριου Κόσα για την πολιτική συνοχής και τις περιφερειοποιημένες κοινότητες. Συμβιβαστική Α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 15. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. Γ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Ι, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, μάλλον όχι, προηγουμένω. Είμαστε στην τροπολογία 13 και θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα ως προσθήκη στο συμβαστικό ε. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτηκε. Να ελέγξουμε. Ωραία, δεύτερο τμήμα της τροπολογία 13. Ψηφίστε. Ψηφίστε. Πέρα τη ε, ψηφοφορία εγκρίθηκε με 29 ψήφου. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε στην τροπολογία 33 το πρώτο τμήμα. Είχε ζητήσει άλλη το ψηφοφορία. Υπέρ, παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16, κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 16 μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις οφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγξουμε. Τροπολογία 21. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε 31 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 26 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 ψήφι υπέρ. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική I υπέρ, κατά, αποχές, ξανά. Συμβιβαστική I, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64. Α, να ελέγξουμε. 62. Τροπολογία 62, έτσι. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα τη Απορρίφθηκε. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροποποιημένη γνωμοδότηση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 42 ψήφοι υπέρ. Και περνάμε τώρα. Ναι. Ναι, ευχαριστώ τον κύριο Κώσα. Ναι. Περάμε στην πρόθεση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. με Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική β, β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την τροπολογία 59. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική D δέλτα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΙΕ. E Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στη σελίδα 8 τώρα, Συμβαστική H, ήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 104, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I, Ι. I, Ι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. να ελέγξουμε. Τροπολογία 13. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική K, κάπα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 39 ψήφοι υπέρ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, συντάκτη την κυρία Γιάννα Σιτνάφσκα. Και περνάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο έκθεσης για τις μονοπρόσωπες εταιρείε περιορισμένης ευθύνης. Να ξεκινήσουμε με τη συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν όλα τα υπόλοιπα και έτσι περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Για το σχέδιο έκθεσης. Το σχέδιο γνωμοδότησης. 35 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Okay, thank you, uh, Madam Steinruck, for this. Σας ευχαριστώ, κυρία Στάινρουκ. Σαφές το αποτέλεσμα. Στο 10 τώρα της μερικής διάταξης. να κάνω μια ανακοίνωση σε σχέση με μια αλλαγή στον κατάλογο ψηφοφορία σε ό,τι αφορά την νομοδότηση του κ. Λόπε. Η τροπολογία υπαριθμών 33 που κατατέθηκε από την κυρία Μαρία Ρένα, Μπαγιέ και Γκουτιέρες Πριάτο δεν ψηφίζεται πλέον ως προσθήκη στην ε, συμβιβαστική ε, θα καταπέσει αν εγκριθεί η συμβιβαστική ε. Και οι προφορικές τροπολογίες έχουν αποσυρθεί πληροφοριακά. Τώρα να ψηφίσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης, για τα Ευρωπαϊκά Δραστηριακά Ταμεία, τα Ταμεία Επενδύσεων και σε ό,τι αφορά τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινωνικών Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε την 19 ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. 30 ψήφι κατά. 21. Υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Και τώρα περνάμε στην συμβαστική ε σελίδα 4 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Α, συγγνώμη, η 43 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. πέρασε. 43 ψήφοι υπέρ. 8 κατά. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στι 3. Ελπίζω, λέει η πρόεδρο, Να είστε εδώ γιατί θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τις συστάσεις χώρα. Τρεις προσκεκλημένους έχουμε, τον κύριο Ντομπρόφσκης, τον κύριο Τέισεν και τον κύριο Μοσκοβισή. Θα προτρέψει η Επιτροπή Οίκων αλλά και η Επιτροπή Απασχόλησης θα συμμετάσχει. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε λοιπόν πάλι στις τρει.